So, ich Παρακαλώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους τώρα να καθίσουν και να ελέγξουν τις ε, κάρτες τους για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Και να αρχίσουμε με την προφορική ερώτηση ΣΥΤΕΣ που ήταν και θέμα σημερινό. Ήταν το 4 και έχουμε την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Παρακαλώ να το υπερψηφίσετε. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με λίγες ψήφους κατά, άρα δεκτό. Θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία, ας το κάνουμε λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ποιο θέμα είναι που ψηφίζουμε, Ρωτάω ο κύριος Ντέιβις είναι το σημείο 4. Για αυτούς τους συναδέλφους που δεν ήταν το πρωί συζητήσαμε το CITES COP16 και επ' αυτού είπαμε ότι θα κάνουμε μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο όμως πρέπει επίσημα, τυπικά, να ψηφίσουμε αυτή την έγκριση για την προφορική ερώτηση. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έλικε η ψηφοφορία. 34 υπέρ, μία, 43 ε, συγγνώμη, υπέρ, μία κατά, μία αποχή.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 65 το πολύ 65, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά. Την 65. Ψηφίσατε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 26 υπέρ. 25 κατά δεκτή. 68 68. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 66, καταπίπτει, 67. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 22, καταπίπτει, 71, έχουμε ξεχωριστεί. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 23, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 70 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας 32 υπέρ 20 κατά μια αποχή ε, εγκρίνεται 75 ε, υπέρ κατά χες, δεκτή. Προφορική τροπολογία Α, καταπίπτει η προφορική τροπολογία και Ψηφίζουμε την 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άφετ 6. Ψηφίζουμε το υπόλοιπο της πρότασης. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σίγουρο, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την ΑΦΕΤ 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 24 κατά, δεκτή. Άφετ 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 77. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 27 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ρέγγι 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ρέγγι 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 34 υπέρ, 22 κατά. Δεκτή. 78 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρί, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, Αποχές. Δεκτή νομίζω, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 84. Ψηφίσατε. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεκτή. 27. Υπέρ. Ρέγγι 27. Υπέρ, κατέ, αποχές, δεκτή. 86. Υπέρ. Ρέγγι Ρέγγι 27 έγινε δεκτή. Δεκτή. Να, να ελέγξουμε παρακαλώ την Ρέγγι, Ρέγγι 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Απορρίπτεται με κάποια πλειοψηφία απορρίπτεται. 86 <laughs> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 89. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Μόνο 20 συνάδελφοι ψήφισαν. 87 ξανά. Υπέρ, κατά, δεκτή. 90 υπέρ, sorry, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91. 91 πίπτη, budget 14, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άθετο 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 95, 96 και άφετε 9 τις ψηφίζουμε όλες μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 80, 98 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 29 υπέρ, κατά, Αποχές. Ε, ηλεκτρονική επιβεβαίωση παρακαλώ. Ψηφίζουμε τη ΡΕΓΚΙ 29. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. 32 υπέρ 29 κατά. Δεκτή. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 ε, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 102 καταπίπτει. 101 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 30. Η επόμενη είναι ΡΕΓΙ 30. Υπέρ. Ρέγγι 30 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται νομίζω λέει ο πρόεδρος. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. 43 υπέρ 19 κατά σαφώ δεκτή 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται 113 υπέρ κατά απόχέ δεκτή Ρέγγι 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ κατά αποχές να ελέγξω ηλεκτρονικά την 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ρέγγι 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 115. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 32. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 116 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, πρώτο τμήμα της 1, ε, συγκεντρωτικής 1. Δεκτή. Πάμε στη ρέγγι 36, υπέρ. Κατά. δεκτή. 37, ε, ρέγγι 37, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Budget 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 dafür. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ενοποιημένη ένα δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά α, αποχές απο, δεκτή δεκτή. Ενοποιημένη ένα. Δεύτερο τμήμα. Ωραία. Προχωρούμε στο άρθρο 7 τροπολογία 144 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 146 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται Regi 44 und Affet 11 werden zusammen abgestimmt. Affet, Affet 11 eh, υπέρ κατά άποχες δεκτή. 145 πρέπει να... Ναι, να την ψηφίσουμε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφε 12. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέγγι 45. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άφε 13. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Ρέγγι 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ κατά 149 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 47 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. ΑΦΕ 14 απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέγγι 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152, 153 ταυτόσιμες και γι' αυτό τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 154 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 154. Ψηφίσατε όλοι, έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 ε, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 155 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 157, 158 ε, ταυτόσημες. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 159 δεν ψηφίζεται. 13, 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 160, 160 δεν ψηφίζονται, τη 17 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 146. 164, συγγνώμη. Απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 167 καταπίπτει. 168 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επιβεβαίωση της 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Ρέγγι 49 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 171 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύε 6 δεν ψηφίζεται. Προχωρούμε στο άρθρο 11, 173 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 174 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 197 υπέρ κατά αποχές δεκτή. άφε 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άφεν 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ Α, ηλεκτρονικός έλεγχος της 179. Ψηφίσατε όλοι, έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Budget 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ντεβε 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε στο άρθρο 13.192. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέγγι 53 υπέρ κατά δεκτή. Budget 20 υπέρ κατά δεκτή. Άφετ 28 υπέρ κατά δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ντεβε 8 και Ρέγγι 54 καταπίπτουν και προχωρούμε 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 28 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 28 παρακαλώ ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία, έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 193. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 194. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε στην 195. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 196. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 δεν πρέπει να την ψηφίσουμε και το 201, 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές δεκτή 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 208 δεν ψηφίζονται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211, όχι, 212 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 210... Α, συγγνώμη, 211 απορρίφθηκε, 212 επίσης απορρίφθηκε, 213 απορρίφθηκε, οι 14, 15, 16 δεν ψηφίζονται, άφετη 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ντεβε 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, άφε 30 υπέρ κατά ε, κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ε, ΑΦΕ 30. Ψηφίσατε όλοι, έληξε ψηφοφορία, απορρίπτεται. 218 δεν ψηφίζεται. 219 την ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, οι δύο επόμενες δεν ψηφίζονται. Άφε 31, ούτε η άφε 31 ούτε 221, ούτε 222, η 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 226 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 227 Πρέπει να ψηφίσουμε την 227 υπέρ κατά Κα... Α, όχι, όχι τη 227, την 31 ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 228, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 229, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Budget 21, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτεται 33 πρώτο τμήμα και εντεύε 11 πρώτο τμήμα ταυτόσημες. Ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ρέγγι 55, Ρέγγι 56 δεν ψηφίζονται. 230 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ελέγχουμε την 33 παρακαλώ, δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή 44 προς 19. Ντέβε Α, όχι. Η 231. Η... Όχι, ούτε αυτή καταπίπτη. 232. Η... 232. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η budget 22. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 233. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 234 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ρέγγι 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή και 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 236 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, 237 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, budget 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 239 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 241 dafür. Dagegen, Enthaltung 241 ε, υπέρ κατά δεκτή, 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 243 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, budget 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 245 υπέρ κατά αποχές ξανά υπέρ τη 245 κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Budget 26 δεκτή. 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 251 καταπίπτει, 256, 200... Αψηφίζονται unblock, 252, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 34, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 256, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ρέγγι 59 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Budget 28. Οι άλλες καταπίπτουν. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 257. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 258. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. ΔΕΒΕ 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 260 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.

αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ τη 263. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις φοφορίες. Σαφώς δεκτή. Αλλά οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες έχουν μια ψήφο παραπάνω. Κάποιος περισσεύει. Ψηφίσουμε. Την 38 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεβε 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 το υπόλοιπο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 κατά πίπτη, 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, άφετ 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 5 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος budget 5. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Πάλι οι σοσιαλιστές έχουν μια ψήφο παραπάνω. Τώρα, τώρα μάλιστα, τώρα είμαστε εντάξει. Έγινε δεκτή. Εν συνεχεία ε, ψηφίζουμε την 48 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ρέγγι 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή Budget 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή Άφετ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέγγι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άφε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέγγι 7 υπέρ κατά Ψηφίζουμε την Ρέγγι 7 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία έλλειξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 3 και ρέγγι 9 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά αποχές, δεκτές. Ρέγγι 8, υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 54, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ρέγγι 10, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Budget 10, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος, budget 10. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. απερίφθη, απερίφθη. Σαφέστατα. Τέσσερα υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Ρέγγι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. steht zur Abstimmung. Dafür? 58 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 3 υπέρ, δεύε 3, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, Ρέγγι 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ρέγγι 16, υπέρ, κατά, α, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος Ρέγγι 16, παρακαλώ. Ε, ψηφίσατε όλοι, έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή, δεκτή. Ε, budget 12 ε, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ρέγγι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. απορύπτετα 4 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άφετ 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 62 κατά καταπίπτει. Ρέγγι 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται η 6 καταπίπτη ρέγγι 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Budget 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αφετ 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, α, απορρίπτεται. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. 52 υπέρ, 5 ψήφοι κατά, 3 αποχές. Συγχαρούμε την συγκίτη, αλλά τώρα πρέπει να ψηφίσουμε και το νομοθετικό ψήφισμα. But Α, συγγνώμη, ένα λεπτό. Budget 2, την budget 2 ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Budget 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία, έληξε ψηφοφορία. 52 ψήφοι υπέρ έναντι πέντε ψήφων και τρεις απόχες. Θερμές χαρητήρια στην κυρία εισηγήτρια, την κυρία Γκαρντίνη. Θέλετε κάτι να πείτε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εποφελούμε τις ευκαιρίες αυτής που μου δίνετε να πάρω το λόγο για να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδης ηγητές για τη συνεργασία τους και θα ήθελα να σας προτείνω να ξεκινήσουμε τις με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας με στόχο να καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση βάσει του άρθρου 70 του κανονισμού μας. Σας προτείνω να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση που μόλις εγκρίναμε ως εντολή διαπραγμάτευσης. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε μια διαπραγματευτική ομάδα όπου η συγκήτρια θα είμαι εγώ, επικεφαλής ο πρόεδρός μας και θα συμμετέχουν βέβαια και όλοι και οι συγκητές. Υπάρχουν αντίρρηση επ' Δεν βλέπω μία αντίρρηση, οπότε έτσι θα προχωρήσουμε με το άρθρο 70. Θα έχουμε ακόμα πολλές ευχάριστες ώρες. Να περάσουμε. Είναι στην ημερήσια διάταξη στις 10 Δεκεμβρίου. Αλλά θα μας δημιουργήσει ακόμα πολλές ευχάριστες στιγμές, όπως σας είπα. Ωραία, εύχομαι κάθε επιτυχία και ολοκλήρωση στην πρώτη ανάγνωση. Πολύ ωραία. Και προχωρούμε στο επόμενο, στην επόμενη ψηφοφορία που είναι οι ουσίες προτεραιότητα στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του κυρίου Ζίμπερ. Και αρχίζουμε. Καταρχάς ενοποιημένη τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το ενοποιημένη 9. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, την ενοποιημένη 8. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Σαφώς. Ε, ενοποιημένη 9, επίσης ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Επίσης απορρίπτεται. Ενοποιημένη 10. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. 45 υπέρ, 14 κατά. Άρα έγινε δεκτή η 10. Υπάρχουν Τίποτα αμφιβολίες, σχόλια. Ωραία. Τώρα προχωρούμε στην τροπολογία 70. Στη σελίδα 6 είναι σε μένα στον κατάλογο ψηφοφορία. Και για να σας ε, ευχαριστήσω όλους, για να σας χαροποιήσω, έχουμε περάσει πέντε σελίδες. Λοιπόν, 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 231 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος στην 72. Ψηφίσατε. Ελέγχουμε την 72. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχουμε την 233. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 75. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη. ψηφοφορία. Δεκτή. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ κατά Ε, να ψηφίσουν ηλεκτρονικά επιβεβαίωση 79 ε, ηλεκτρονικά υπέρ, κατά, ε, συγγνώμη, έληξε ψηφοφορία, α, απερίφθη. 80 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 235 υπέρ κατά να ελέγξω ηλεκτρονικά 235 ψηφίσατε έληξε ψηφοφορία απορρίπτεται ενοποιημένη 4 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 237 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ένα λεπτό λέει ο πρόεδρος. 237 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 93. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 238 υπέρ 238 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 94 αποσύρθηκε, 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή 240 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση της 12. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές δεκτός. Προχωρούμε στη σελίδα 13, 156, Ούλμερ, 156, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20, 251, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 252 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23-159 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Να ελέγξουμε την 23 και 159 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Ξανά, επαναλαμβάνουμε, 24, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Έχουμε τώρα μία διαχωρισμένη ψηφοφορία για την 32. Ε, να ελέγξω ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. Δεκτή. Α. Ναι, δεκτή με ζάλισε ο Chris Davis και είπα απορρίπτεται. Α, τώρα προχωρούμε στα δύο τμήματα της 32. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελειώνει 38 υπέρ 35 Α, καταπίπτει 35 η 30 έγινε δεκτή. Άρα καταπίπτει 35. Προχωρούμε. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ένα ποιημένη. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε ε, την 49 ηλεκτρονικός έλαχος. ψηφίσατε ε, τέλος της οφορίας Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη. 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να, ηλεκτρονικό έλεγχος. Γιατί πολύ λίγοι ψήφισαν. Λοιπόν, να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Ορίστε. Δεκτή. Σηκώστε το χέρι σας. Τα γέλια δεν ωφελούν. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ως συνένεση και υπερψήφιση το γέλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. 54. Ο κύριος Ζήμπερ. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ. Την τρία. Την τρία που είναι δική μου του εισηγητού. Λοιπόν, α, α, απερίφθη η τρία λέει ο πρόεδρος, αλλά ας ξανα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 3. Ψηφίσατε. Έληξε η ψηφοφορία. Απερίφθη η 3. Προχωρούμε στο 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57. Υπέρ. 55. Πρέπει να ψηφίζουμε την 55. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ και 67 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ ψηφίσατε όλοι την 66-67 έληξε ψηφοφορία δεκτές 68 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 69 Είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο. άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. 64 46 υπέρ, 7 κατά, 6 αποχές. Έγινε δεκτή το σχέδιο έκθεση και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία με 43 υπέρ 7 κατά δεκτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ Ρίχακ και θερμά συγχαρητήρια. Ο Ρίχαρτ Ζίμπερ. Θέλει να μιλήσει για το άρθρο 70. Όπως και η συνάδελφος κυρία Γκαρντίνη, θα ήθελα να συνεργαστούμε όλοι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση βάσει του κανόνα 70 για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις διαβουλεύσεις ε, με το Συμβούλιο και θα πρέπει οι εισηγητές να συμμετάσχουν και σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα μας ενημερώνουν τακτικά. Αυτή, αυτό το αποτέλεσμα της ισοφορίας αποτελεί μια καλή βάση για την περαιτέρω διαπραγμάτευση. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Δεν νομίζω. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, το θέμα είναι θέλουμε να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση. Αν θα δοθεί εντολή ή όχι. Τι θέλετε να κάνουμε. Να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την πρόταση συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. 44 υπέρ 7 κατά 2 αποχές. Άρα υπάρχει εντολή, δίνουμε την εντολή για μια συμφωνία προς την πρώτη ανάγνωση. Ωραία. Εξασκούμε τώρα, εφαρμόζουμε την νέα ερμηνεία του κανονισμού. Έχουμε ήδη τεράστια αύξηση του ποσοστού συμφωνίας ε, στην πρώτη ανάγνωση. Είναι μια τεράστια αύξηση αυτού του ποσοστού και είναι μια πολύ καλό γεγονός. Ε, να προσθέσω ακόμα, αλλά ε, όλοι ξέρετε τι συμφωνήσατε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, ότι το θα, ψηφίσετε εδώ στην Επιτροπή και για το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για ένα ναι ή ένα όχι. Όπως σας είπα, θα περάσουμε ευχάριστες ώρες και δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Προχωρούμε στο 13, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις είναι του κυρίου Χρυσόγελου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Την είχαμε αναβάλει, έγινε περαιτέρω επεξεργασία και αρχίζουμε κατευθείαν. Υπάρχουν τίποτα παρατηρήσεις, απορίες. Όχι. Ωραία. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 138. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. 172 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 172. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και τροπολογία τρία, Πέρας. Απορρίπτεται. Οι 173-176 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 174 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Περνάμε στην 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Έλεγχος. Για την 8, ναι. Ελέγχουμε για την τροπολογία 8, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Επρόκειτο για ομαδοποιημένη μας τροπολογία. 206 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ομαδοποιημένη 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 221 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 268 υπέρ κατά απορρίπτεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε για αυτή την τροπολογία 277 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά. Για 279 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 280 υπέρ. Μάλλον κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για 279 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 290 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού ψηφίζουμε τις 293 945 υπέρ κατά εγκρίνονται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ομαδοποιημένη 23 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Σαρανταπέντε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 305 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 306 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 307 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 308 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 309 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 313 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 314 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά 321 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 και 323 είναι ταυτόσιμες, από κοινού ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 324, κατά, απορρίπτεται, 325 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51. Θα κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική επαλήθευση για την 326 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 327 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 328 άρτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 332 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 332 σας παρακαλώ, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 333 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ κα, μάλλον πίπτη. 336 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 337 υπέρ κατά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 εγκρίνεται 348 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 349 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 350 υπέρ, κατά αποχές Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για 350 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 351 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 352 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 354 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 355 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 356 υπέρ κατά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 δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. 362. Συγγνώμη, καταπίπτει. 363 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 363 παρακαλώ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οματοποιημένη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 371 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ομαδοποιημένη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θα κάνουμε έναν, μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την 75, σας παρακαλώ. Άρτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την ομαδοποιημένη 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ομαδοποιημένοι 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ, καταπίπτει 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 104. Πέρας. Εγκρίνεται 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 110. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114, 115 ταυτόσιμες, επομένως από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 114 και 115. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 44 υπέρ εγκρίνονται λοιπόν. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 118. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται, 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είχαμε πολλές ηλεκτρονικές ψήφους, ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση αυτή. Πέρας. 49 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Ωραία, προχωράμε τώρα στο θέμα του αμίαντου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Βίλς και αρχίζουμε αμέσως με τις... Συγγνώμη, είπε ο πρόεδρος. Σιγά σιγά, να πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, έχουμε την τροπολογία 1 υπέρ του τίτλου κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, ενοποιημένη 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τελειώνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι έληξε ψηφοφορία 49 προς ψήφο, καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Βίλς. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες και μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα 15. Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζει στη μέση των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστου στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας. Προτείνω να δώσουμε την ευκαιρία σε όσους θέλουν να μείνουν, να μείνουν και όσοι δεν επισημούν να συνεχίσουν στη συζήτηση να μείνουν, να φύγουν από την αίθουσα ήσυχα και ωραία. Ωραία. Δίνω καταρχάς το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία. Ησυχία στην αίθουσα για να μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Παρβάνοβα, η οποία έχει το λόγο. Bitte, Frau Η κυρία Παρβάνοβα. Πρόεδρε, για όλου του συναδέλφου που έχουν υποβάλει τροπολογίε και έχουν κάνει προτάσει για φωτοζωτική σημασία και πολύ ευαίσθητο θέμα, ότι του ευχαριστώ ιδίω του κοιόδη συζητητέ για την καλή συνεργασία και την προθυμία του να έχουμε διάλογο και να βρούμε ε, σταθερέ και αποτελεσματικέ συμβαστικέ λύσει. Εργαστήκαμε πολλέ πλειά στι συναντήσει με του κοιόδη συζητητέ για τον σκοπό αυτό και τώρα θα θέλω να παρουσιάσω τον καρπό των έργων μα και να σταθώ στα σημαντικότερα σημεία όπου προσπαθούμε να βρούμε μια τοποθέτηση αποδεκτή από όλου. Αναζητούμε το, ε, ένα σύνολο συμβαστικών προτάσεων, ενό τέσσερα, για τις αποφάσει τιμολόγηση και επιστροφή δαπανών και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πάμε προς την εξή κατεύθυνση. Ε, διαγραφή της διτής χρονική γραμμή για τα φάρμακα που διαθέτουν ε, την άδεια HTA, 90 ημέρες για την επιστροφή, 180 και 90 για την τιμολόγηση και 90 για την επιστροφή, 180 συνολικά, μία και μόνη γραμμή για τα γενώσιμα, 30 για την τιμολόγηση και 30 για την επιστροφή, 60 συνολικά. Και τέλος, αναφορά στην αποτίμηση των ε, απαιτήσεων υγεία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόσουν τις σχετικές υποχρεώσεις, ε, η χρονική αυτή γραμμή θα πρέπει να θεωρηθεί απόφαση των αρμοδίων αρχών, αλλά με μία ενιαία χρονική γραμμή. Μια άλλη συμβαστική λύση, η 5, αφορά το άρθρο 8. Προβλέπει τα ένδικα μέσα εδώ θέλουμε να γίνει πιο ήπια η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μιλώντας για διαμεσολάβηση και διαδικασίες προσφυγής, ώστε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν πώς θα διασφαλίζουν την ε, παροχή ε, ένδικων μέσων και δυνατότητας διαμεσολάβησης. Έπειτα, για το άρθρο 13 και τις πρόσθετες αποδείξεις για την ποιότητα και την ασφάλεια και την βιομοιότητα, εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί η πρόταση της Επιτροπής με επικεντρωνόμενη σε μία βασική αρχή. Τα στοιχεία της ε, αδειοδότησης. Επίσης, θέλουμε να εγγυηθούμε ότι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της διαδικασίας ε, αδειοδότησης για εμπορία και της τιμολόγησης και επιστροφή δαπανών δεν πλήττει τις εθνικές αρχές στις υποχρεώσεις τους για την συγκέντρωση στοιχείων και πρόσθετων δεδομένων. Επίσης, αναζητούμε συμβαστική λύση για να ενισχύσουμε την αρχή της διαφάνειας με τη συμβαστική λύση 7 συγκεκριμένα, προσπαθώντας να επικεντρώσουμε σε βασικούς τομείς όπως τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων και τη δήλωση συμφερόντων τους, την ε, υποχρέωση αποκάλυψης του απορρίτου σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται και επίσης την κοινοποίηση των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε άλλα τμήματα του κειμένου Υπήρξαν και άλλε τροπολογίε από του συναδέλφου και ευχαρίστως να ακούσω τις απόψει τους εδώ. Απλώς να αναφέρω μια διάταξη που θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει συνεπής και αντικειμενική. Το άρθρο 14. Την μην ε, παρεμβολή των δικαιωμάτων πνευματικη ιδιοκτησια Η σχετική πρόταση τη ευρωπαικη επιτροπη είναι μια ε, μετάφραση, πιστή μετάφραση των συστάσεων του 2007 που προέκυψε από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Εντοπίστηκαν εδώ πρακτικές ε, στρεβλωτικές του ανταγωνισμού σε σχέση με την διάθεση στην αγορά γενώσιμων προϊόντων τα οποία μας μπορούν να επιτρέψουν και εξοικονόμηση στα δημόσια συστήματα υγείας. Δεν βλέπω λοιπόν εδώ βάσιμους και αντικειμενικούς λόγους να ξανανοίξει το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το άρθρο 14 θα πρέπει να μείνει όσο έχει και όσο έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει τη σχετική μελέτη. Επίσης θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι και τι μπορεί να συμβεί στο Συμβούλιο, διότι όπω τα γνωρίζουν και οι συνάδελφοι στο Κοινοβουλίο, υπάρχει και κάποια σχετική πρόοδο στο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση. Προφανώς είναι δύσκολο να συνεχίσει να αποτελεσματική μια 20 οδηγία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσει για την επιστροφή δαπανών είναι σαφεί για όλου, ότι είναι διαφανεί, ε, βασίζονται σε συγκεκριμένα αποδεκτικά στοιχεία και επιτρέπουν την πραγματική πρόσβαση των ασθενών σε νέε και σε λογικές τιμές ε, φαρμακευτικές αγωγές. Τροποποιήσαμε την αρχική ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο χρονικό της όριο, αντιμετωπίσαμε και συγκεκριμένε μέρημνες των κρατών μελών και των εθνικών αρχών και νομίζω ότι αυτή η επικοδομητική προσέγγιση πρέπει να συνεχιστεί. Να εξεύρουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η συγγήτρια του ΕΛΚ, η κυρία Ρούκοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους ισχυώδεις εισηγητές, διότι η εργασία που έκαναν ήταν εξαιρετική, ομαδική εργασία. Ξέρω ότι πολλά κράτη ε, έχω προβλήματα με αυτή την οδηγία. Αλλά η συμφωνία είναι ουσιαστική, ουσιώδου σημασία και προσπαθούμε ακόμα περισσότερο να κάνουμε ρεαλιστική την οδηγία. Πρέπει να υιοθετήσουμε νέα μέτρα και να έχουμε υπόψη τους ασθενείς μας για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή τους μεταχείριση. Πέραν αυτού, το θέμα της διαφάνειας σε αυτό τον τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι είναι ουσιαστική σημασία και για τον τομέα και για τα κράτη-μέλη. Το ΕΛΚ έχει υποβάλει τροπολογίες και συμβιβαστικέ τροπολογίες ε, με ουσιαστικό περιεχόμενο. Έχουμε υποβάλει προτάσεις για νέα ε, χρονοδιαγράμματα και επίσης ε, καταφέραμε να, να συμφωνήσουμε επί του άρθρου 8 έχουμε, δεν έχουμε διαγράψει όλο το άρθρο, αλλά έχουμε αφήσει δύο πιο ήπιες παραγράφους. Με τις τροπολογίες μας, επίσης, καταφέραμε να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να έχουν πλήρη πρόσβαση ε, στα δεδομένα, στα στοιχεία και να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης πρόσθετων στοιχείων. If orphan ότι θα πρέπει να προληφθούν και τα ορφανά at our group. διότι αυτό το έχουμε συζητήσει στην ομάδα μας. Πράγματι υποστηρίζουμε την διαφάνεια, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όμως υπάρχουν ακόμα ορισμένοι ορισμοί που πρέπει να διευκρινιστούν. Έχουμε ακόμα ε, λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για περισσότερες διαβουλεύσεις και πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό. Παρακαλώ, ε, μελετήστε, ο, μελετήστε όλα τα, τις πτυχές και υποστηρίξτε τις τροπολογίες μας. Ο πρόεδρος, η συγγήτρια από τη σοσιαλιστική ομάδα και δημοκρατική ομάδα. Ευχαριστώ πρόεδρε, η κυρία Τσίλτερς. Είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας μεταξύ των κρατών μελών και άπτεται των εθνικών συστημάτων υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανία και της πρόσθετης αξίας την οποία μπορεί να προσδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ασθενείς. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία μαζί μου. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες αυτές για να καταφέρουμε να περιορίσουμε το διοικητικό άχθο στα κράτη-μέλη και να μην δυσκολέψουμε τις αποφάσεις για την τιμολόγηση. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για να μειώσουμε τα άρθρα που αφορούν ε, τις κυρώσεις και τα ένδικα μέτρα. Επίσης ε, μέτρα για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά των γενώσιμων φαρμάκων και διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων. Θα εξετάσουμε λοιπόν από κοντά όλες τις τροπολογίες για να δούμε εάν διευκολύνουν και ενισχύουν την διαφάνεια ε, και λαμβάνουμε υπόψη και τις επιφυλάξεις όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρμοδίων αρχών. Επίσης, ε, ήδη χρησιμοποιείται η, η, η, η βάση δεδομένων Euripid από 20 κράτη-μέλη η οποία προσφέρει και αυτή ορισμένες διευκολύνσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα. Δεν είναι δημόσια αυτή η βάση δεδομένων, χρησιμοποιείται όμως από τα, από τα κράτη-μέλη. 150.000 ευρώ το χρόνο κοστίζει η λειτουργία και πιστεύω ότι αξίζει να τη διατηρήσουμε όπως έχουμε υποβάλει τροπολογία 259. Έχουμε λοιπόν υποβάλει τροπολογίες και συμβαστικές τροπολογίες που εκφράζουν τις απόψεις μας. Ευχαριστώ. Εν συνεχεία. Εκπρόσωπος των Πρασίνων, υπάρχει κανείς? Όχι. Για την... Αλτα Σούσα, το Κυρία Σούζα. Όχι. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι κράτη-μέλη ήδη δυσκολεύονται να ισοσκελίσουν ε, τα δημοσιονομικά τους και πρόθεσμα και να καλύψουν τα, τις δαπάνες των φαρμακευτικών προϊόντων. Νομίζω λοιπόν να θεωρήσει τις οδηγίες αυτής για την διαφάνεια θα πρέπει να εξετάσει και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις επιδόσεις καινοτομία και τεχνολογικές ε, επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υγειονομική ασφάλεια μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουμε μια σαφή μερίμνα και να βρούμε τη σωστή ισορροπία της ε, αποζημίωσης της ε, αμοιβή για την ε, καινοτομία, της καλής πρόσβασης στα φάρμακα και την ε, διατήρηση του εύλογου κόστου των συστημάτων κοινωνική πρόνοιας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών των φαρμάκων χωρίς να ξαναδούμε το όλο σύστημα διοδότησης των φαρμάκων που ορίζεται από την Οδηγία 2003 για την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος. Το κείμενο αυτό έχω υποβάλει και εγώ κάποιε τοπολογίε διότι ήθελα να σταθούμε στο ότι δεν πρέπει σε εθνικό επίπεδο να εξετάζουμε την ιατρική ε, προστιθέμενη αξία των ορφανών φαρμάκων. Εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη η υγειονομική περίθαλψη είναι αρμοδιότητα εθνική, αλλά κάποιες φορές περιφερειακή ή και τοπική. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε την περιττή ε, των ε, χρονικών προθεσμιών και του διοικητικού κόστου. Θα πρέπει και οι διοικητικές αρχές να φροντίσουν να μην υπάρξει αντίκτυπο στι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διαδικασίες. Έχω λοιπόν υποβάλει σχετικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα έχει το λόγο. Α, κύριε Έμπνερ, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίμπνερ είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική ε, διάταξη αυτή ε, για το πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει ένα φάρμακο στην αγορά. Αυτό δεν έχει μόνο επιπτώσει στην υγεία και στη ζωή των ασθενών, αλλά η κυκλοφορία ενός φαρμάκου έχει σαφώς επιπτώσεις και στους κατασκευαστές. Μπορεί, στους παρασκευαστές, μπορεί κάποια στιγμή να αποδειχθεί ότι όλη η διαδικασία είναι προβολικά χρονοβόρα. Η επιτάχυση αυτής της διαδικασίας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην αγορά. Παλιότερα οι πληροφορίες που είχαμε για τα φάρμακα ε, ήταν διαθέσιμες στα ειδικά, στις ειδικές εκδόσεις περιοδικά και φυλάδια του τομέα. Τώρα όμως ε, δίνουμε το δικαίωμα και μέσω του διαδικτύου κάθε πολίτης να μπορεί να εξετάσει τις ιδιότητες των, ενός φαρμάκου, αν μπορεί να το αγοράσει, πού και πώς και αν είναι διαθέσιμο στην αγορά. Για τους ασθενείς αυτή η διαενημέρωση, αυτές οι πληροφορίες έχουν μεγάλη, τεράστια σημασία. Είναι σαφές ότι μέσα στα ασφαλιστικά ταμεία τώρα έχουμε πάρα μεγάλες περικοπές και θα πρέπει να επαναφέρουμε ε, μία ισορροπία στο πλαίσιο των συστημάτων ασφάλισης υγείας. Η Επιτροπή τώρα. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια πρόταση αρκετά δύσκολη. Αυτή παράδοση τη χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο, τους εισηγητές και την κυρία Παρβάνοβα για τις προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Νομίζουμε ότι υπάρχει καλή προαίρεση και καλό πνεύμα συνεργασία για να ολοκληρωθεί το όλο θέμα και σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την πραγματιστική και ευέλικτη προσέγγιση που έχει ακολουθήσει ω τώρα στι διαπραγματεύσει προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αίσιο πέρα. Βεβαίω θα πρέπει να βελτιωθεί η ισχύουσα κατάσταση σε σχέση με την ε, ισχύουσα νομοθεσία και οδηγία. Οπότε πρόθεσή μας δεν είναι να οπισθοχωρήσουμε, αλλά να προοδεύσουμε σε αυτή τη φάση απλώς να εκφράσω την ε, εμπιστοσύνη μου στην ε, μελλοντική καλή συνεργασία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ώστε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε και την Κυπριακή Προεδρία για τις όλες τις προσπάθειες και ελπίζουμε στην πλήρη συνεργασία της Ιρλανδικής Προεδρίας που έπεται. Ελπίζουμε ότι θα επιτελέσουμε πρόοδο και επιτρέψτε μου να πω ότι η σημερινή συζήτηση είναι ένα πολύ θετικό δείγμα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ευχαριστώ και δίνω ξανά το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ και πάλι. Δηλώνω ότι είμαι αποφασισμένη να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά για το θέμα αυτό, σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητέ και σε όλο αυτό το θετικό πνεύμα. Όλοι συμπλέουμε στο στόχο μας Έχουμε μια κοινή θεώρηση του θέματος γιατί μας απασχολούν και η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και οι καινοτόμες θεραπευτικές αγωγές και η ασφάλεια προς όφελος των καταναλωτών, αλλά και η δημοσιονομική σταθερότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας. Υπάρχουν κάποια κρατημέλη που ίσως έχουν ακόμη επιφυλάξεις, αλλά να αποστείλω το μήνυμα από την πλευρά όλων των σκιωδών ότι πραγματικά λαμβάνουμε υπόψη τις πιέσεις, τις δυσκολίες, τους τριγμούς που αυτή τη στιγμή γνωρίζουν. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή τους και για όσους έχουν κάποια τοποθέτηση σε εθνικό επίπεδο με αφορμή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πούμε ότι φροντίσαμε να ε, προσαρμοστεί πάρα πολύ η πρότασή μας ώστε να προσεγγίζει αυτή του Συμβουλίου. Πραγματικά ελπίζουμε στην καλή μας συνεργασία και ελπίζουμε να περατωθεί πολύ γρήγορα το ευαίσθητο αυτό νομοθέτημα στην εξέτασή του. Με τρόπο πραγματικά επιτυχημένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Την Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 19 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε και δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για την Ολομέλεια. Επόμενο θέμα είναι το 16, τροποποίηση της οδηγίας 2006-66 για τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στυλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για σύρματα ηλεκτρικά εργαλεία. Εδώ ο κύριος Παναγιώτοφ είναι εισηγητής και θα του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πολύ σημαντική αυτή οδηγία που έχει να κάνει με τις ηλεκτρικές στήλες και τους ερευτές που περιέχουν κάδμιο. Θα είμαι σύντομος και θα ήθελα να μιλήσω όμως τη γλώσσα μου, τα βουλγαρικά. Η οδηγία 2006 66 αναφέρεται στους ε, ε, φορητούς ηλεκτρικούς στις φορητές ηλεκτρικές στήλες που έχουν πάνω από 0,002% κάδμιο. Και υπάρχουν εξαιρέσεις βεβαίως, γίνονται εξαιρέσεις ε, για συναγερμούς και ε, ε, φωτισμούς έκδετης ανάγκης, ειδικού εξοπλισμού και ασύρματα ηλεκτρονικά εργαλεία. Υπάρχουν ορισμένε εξαιρέσει γι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε αυτή τη διαδικασία τώρα. Επειδή εμπλέκονται επικίνδυνε ουσίε και μάλιστα χημικέ ουσίε και επειδή το κάδμιο είναι βλαπτική ουσία, και έχει βλαπτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Το καδμίο είναι τοξικό σε πυκνότητα όταν υπάρχει στο περιβάλλον και το κάδμιο μπορεί επίσης να ε, δημιουργήσει μη αναστρέψιμες βλάβες. Θέλω να παρατηρήσω ότι εάν έχουμε σωστά συστήματα ανακύκλωσης και εάν έχουμε μία σωστή λειτουργία των φορητών ηλεκτρικών συσκευών ε, με τα σωστά συστατικά, τότε μπορούμε να επιτύχουμε μία μη βλαπτική ανακύκλωση και μπορούμε να ακυρώσουμε και να ξεπεράσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο για το περιβάλλον και στους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε δηλαδή 100% να ανακυκλώσουμε αυτές τις, ε, αυτά τα εργαλεία, τα ηλεκτρικά εργαλεία εφόσον χρησιμοποιούμε ε, ιόντα λυσίου. Αυτές οι μπαταρίες ε, λυσίου, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις ε, μπαταρίες νικελίου, καδμίου, νικελίου, μεταλλίου, θα κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, είναι πιο αποτελεσματικές σε αποπόψεις κατανάλωσης ενέργειας, αλλά έχουν λιγότερο διάρκεια ζωής. Επίσης δεν λειτουργούν ε, πολύ καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν επαρκή οικονομικά κίνητρα για τη χρησιμοποίησή τους σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, παρατείνουμε την ρήτρα εξαίρεσης για ένα χρόνο ακόμα, από 31 12 ε, ε, του 11 μέχρι 31 12 του 2016 για άλλο ένα έτος μέχρι το τέλος του 2016 γιατί αυτό θα αποτελέσει μια λογική συμβαστική λύση θα, συμφε... θα προστατεύσει και τους καταναλωτές και τους επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις και ε, επίσης ε, δεν θα βλάψει ούτε το περιβάλλον ούτε την ανθρώπινη οδηγία ενώ ταυτόχρονα θα παράσχει πρόσθετο χρόνο για τεχνολογικές εξελίσεις ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτομίες πολλές ε, φορές τίθεται το ερώτημα πώς κατασκευάστηκαν αυτά τα προϊόντα ε, που βρίσκονται στην αγορά εφόσον ήδη υπάρχει αυτή η απογόρευση και επίσης τα ανταλλακτικά. Ε, πρέπει να πληροφορήσουμε τους ε, ε, ε, κατασκευαστές πότε θα ισχύσει αυτή η απαγόρευση και μετά, να τους πούμε ότι μετά από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν αυτό στις μπαταρίες νικελίου καδμίου, νικελίου μεταλλίου. Νικελίου μετάλλου, συγγνώμη. Θα υπάρχει οριστική πάυση αυτών των μπαταριών. Επίσης, αν δούμε τώρα την οδηγία και αν την επεξεργαστούμε εκ νέου, θα πρέπει να τονίσουμε και επίση το πρόβλημα της ελευθέρωσης υδραργύρου στο περιβάλλον. Γι' αυτό προτείνω στις 31 Δεκεμβρίου 2016 να απογορευτεί η χρήση μηχανημάτων που περιέχουν υδράγυρο ο οποίος μπορεί να ελευθερωθεί στο περιβάλλον. Ε, ιδίως ε, στους παραγωγούς στοιχείων κουμπιών που πρέπει να αλλάξουν την τεχνολογία αυτή. Εάν δεν γίνει αυτή η αλλαγή, τότε θα είχαμε 2,5 με 4 τόνους τριεργύρου ετησίως, ε, ένα πάρα πολύ βλαβερό στοιχείο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ορισμένε πολιτείε των ΗΠΑ έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση στοιχείων κουμπιών με υδράργυρο. Γι' αυτό λοιπόν και από ό,τι προκύπτει από την ε, συνθήκη της Λισαβόνα, ε, πρέπει να, να μειώσουμε τις μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις ε, στο ρήπανση με τον υδράργυρο και να λάβουμε υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα και στην οδηγία αυτή και για τις στήλες ε, και για τη μείωση των βλαπτικών επιπτώσεων. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή. Ξέρουμε όμως είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε αυτά τα ζητήματα και για να πετύχουμε και πλήρη διαφάνεια και ε, σαφήνεια ε, πιστεύω ότι θα πρέπει η Επιτροπή μας να κάνει μία γνωμοδότηση όσον αφορά τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν επ' αυτού τα μέλη μας. Και τέλος προτείνω μέχρι τις 31 Δεκάτου 2006 ε, να παρατείνουμε την ε, ρήτρα εξαίρεσης για να μπορέσουμε εν τέλει να επιτύχουμε την ανακύκλωση σε ποσοστό 100% την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στο, όταν υπάρχει κάδμιο στις ηλεκτρικές στήλες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή, αυτός ο συμβασμός θα έχει θετικά αποτελέσματα και θα εξυπηρετήσει και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στη σκιώδη συγγήτρια, την κυρία Κούκοβιτς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όχι μόνο για το έργο του, αλλά και για τις διαβουλεύσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα συμφωνήσω με κάποιες τις τροπολογίες που προτείνει, αλλά όχι με το σύνολό τους. Θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και εντός του ΕΛΚ, ώστε να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε περιβαλλοντικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις από τις αλλαγές ε, που θα προκύψουν με την οδηγία. Η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες ουσιαστικά έχει ένα λεπτομερή κατάλογο εξαιρέσεων ε, και σχετικά κριτήρια. Οι αλλαγές όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οδηγία με σκοπό να αλλάξουν μόνο οι Διατάξει για τους συσσωρευτέ και τις ηλεκτρικέ πύλες νικολίου καδμίου είναι μια απαραίτητη επικαιροποίηση. Όμως, το σύνολο της πρόταση τη Επιτροπή επικεντρώνεται μόνο σε αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο και η μελέτη αντικτύπου μελέτησε τη συγκεκριμένη και μόνον εξαίρεση και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την οικονομία. Ο εισηγητής στα πλαίσια του έκθεσή του, ε, έλαβε υπόψη και τα στοιχεία κουμπιά που συμπεριλαμβάνουν υδράργυρο, διευρύνοντα το εύρο τη εξέταση του θέματο. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την ανθρωπινή υγεία, όπω και τα παιδικά παιχνίδια. Είναι από τα βασικά ε, προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία κουμπιά. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί τα παιδιά πλήττονται κυρίω από τα ποσοστά για τι συγκεντρώσει υδρακύρου. Πρέπει λοιπόν οι ίδιε διαδικασίε που έγιναν για την ε, μελέτη του, του αντικτύπου νικελίου καδμίου να γίνει και για τα στοιχεία κουμπιά, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε την ε, περίπτωση προσαρμογής και αλλαγής όπως θα γίνει με την απαγόρευση του καδμίου. Ε, εγώ πιστεύω ότι και για, τη, για όλες τις περιβαλλοντικά επιζήμιες ουσίες πρέπει να υπάρξει παρόμοια διαδικασία. Στα ίδια χρονικά πλαίσια. Βεβαίω με κάθε απαραίτητη κοινή λογική. Η όλη διαδικασία ανακύκλωση των ηλεκτρικών στυλών καδμίου, ε, των νέων μάλλον ε, στυλών θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει δικού της πόρους και τις πραγματικές της πρώτες ύλες η Ευρώπη. Θα πρέπει ε, να συγκεντρώνουμε και να αξιοποιούμε αυτά που ήδη διαθέτουμε με τρόπους που να είναι περιβαλλοντικά ασφαλείς και να τονώνουν την οικονομία μας. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω τη στήριξή σας για τις τροπολογίες μας που θα προκύψουν στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστώ. Τώρα συγγητής από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας θυμίσω λίγο γιατί μιλάμε εδώ. Το κάδμιο είναι μια πολύ επικίνδυνη ουσία. Στον κανονισμό REACH έχει κατηγοριοποιηθεί ως κατηγορία η οποία προκαλεί πάρα πολύ σημαντικές ανησυχίες. Βέβαια, αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ουσία αυτή είναι τοξική για τους ανθρώπους και καταστρέφει το περιβάλλον. Ξέρετε ότι λάβαμε υπόψη μας την πληροφορία αυτή στον κανονισμό που είχαμε και το 2006. Ο λόγος όμως για τον οποίο δεν, δεν συμπεριλάβαμε τότε τις ηλεκτρικές στήλες ήταν επειδή περισσότεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσαμε ότι ε, υπήρχαν εναλλακτικέ λύσεις στον βιομηχανικό αυτό κλάδο. Μάλλον, λέγαμε τότε ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικέ. Ξέρουμε όμως ότι τώρα υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις και θα μπορούσαμε αυτές να προωθήσουμε. Συνήθως όταν ε, νομοθετούμε για τις χημικές ουσίες, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλήξουμε σε κανονισμούς οι οποίοι προωθούν την καινοτομία. Θα θέλαμε δηλαδή να βοηθήσουμε προφανώς την προστασία του περιβάλλοντος και να διασώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αν περιμένουμε μέχρι οι δυνάμεις της αγοράς να επιφέρουν τις αλλαγές αυτές, τότε για ποιο λόγο να νομοθετούμε, είναι εντελώς περιττό. Αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνουν πιο φθηνές οι ηλεκτρικές στήλες καδμίου, τότε για ποιο λόγο εμείς να νομοθετούμε τώρα. Νομοθετούμε όμως ακριβώς επειδή θέλουμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και αυτό έχουμε κάνει και με πάρα πολλά άλλα θέματα και κάτι τέτοιο ακριβώς θα πρέπει να πράξουμε και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σας προκαλεί λοιπόν εντύπωση το ότι δεν συμφωνώ με τον εισηγητή όταν λέει ότι θα πρέπει να παρατείνουμε την προθεσμία από το 2016 στο 2017. Αντίθετα, εγώ θα έλεγα να φέρουμε στο 2014, πιο νωρί την καταληκτική ημερομηνία απόσυρση ε, των ουσιών αυτών. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έχει κάνει πραγματικά μια εξαιρετική εργασία. Η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή σε πάρα πολλά σημεία. Μ' αρέσει επίση πάρα πολύ το γεγονό ότι θέλετε να συμπεριλάβετε τον υδράργυρο που εμφανίζεται στα στοιχεία κουμπιά. Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Μολονότι πιστεύω ότι όπω και με το Κάθμιο δεν υπάρχει κανένα λόγο να προβλέπετε μια αναβολή τη προ... προθεσμία ω το 2017. Θα πρότεινα και για τον υδράργυρο ω καταληκτική προθεσμία το 2014 και ελπίζω να υποστηρίξετε την πρότασή μου αυτή όταν θα περάσουμε στι διαπραγματεύσει. Νομίζω πίσω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο εισηγητή προτείνει όλες οι ηλεκτρικές στήλε και σωρευτές με κάδμιο, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία κουμπιά με υδράργυρο, θα πρέπει να αποσυρθούν εντελώς από την αγορά όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία. Όχι μόνο δηλαδή να μην υπάρχουν νέα τέτοια προϊόντα στην αγορά, αλλά να αποσυρθούν και τα υφιστάμενα προϊόντα κατά εκείνη τη χρονική στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργενσεν. Ο κύριος Καρλ Λούτενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Γιούλιος, είσαι πολύ άτυχος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε ένα νέο μέτρο όπου να επιβάλλεται μία απόσυρση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην προβλέπεται μία επιμέρους απόσυρση από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε μάλιστα να μειώσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα ποσοστά 5, 10, 15% ακριβώς επειδή δεν έχουν κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν. Στο άρθρο 11 λέγεται ξεκάθαρα ότι ε, ε, οι ηλεκτρικές στήλες θα πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται από τις διάφορες συσκευές. Όλοι μπροστά σας, για παράδειγμα, έχετε μία μικρή οθόνη, στην οποία βέβαια είναι αδύνατο να αφαιρεθεί η μπαταρία, η ηλεκτρική στήλη. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί παραβίαση της σχετικής οδηγίας και δεν θα έπρεπε να γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι πολύ επικίνδυνο για το περιβάλλον το φαινόμενο αυτό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την μπαταρία από τις συσκευέ αυτές και πολλές φορές χρειαζόμαστε να αγοράσουμε μία νέα συσκευή. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11. Επίσης, δεν προβλέπεται μία εξαίρεση από την αποθήκευση των δεδομένων όπως θα έπρεπε να γίνεται εδώ πέρα. 2009 επίσης, το 2009 ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να είχε υποβάλει μία πρόταση όσον αφορά την σήμανση για την ικανότητα και πάλι εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο ήταν ένα από του πιο σημαντικού αγώνε που είχαμε δώσει στο παρελθόν, όπου είχαμε επιμείνει ακριβώ τα δύο αυτά ζητήματα. Είχαμε πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο τέλο των διαπραγματεύσεων αυτών τελικά συμφωνήσαμε ότι το 2009 θα είχαμε capacity labeling για τι μπαταρίε μια χρήσεως, τι ηλεκτρικέ στήλε μια χρήσεως, καθώ επίση και για τι ηλεκτρικέ στήλε, οι οποίε είναι ενσωματωμένε μέσα σε συσκευέ. Και είχαμε πει πάλι τότε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλαμε μια συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία συμπεριλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στο άρθρο 11, το οποίο στην πράξη όμω δεν έχει εφαρμοστεί. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καλύψετε αυτέ τι αδυναμίε. Τώρα να έλθω στην έκθεση του εισηγητή. Το 2006, όταν διαπραγματεύτηκα το ζήτημα αυτό, είχα κάποιους που ήταν από τη μία πλευρά και από την άλλη κάποιου άλλου που ήταν από την άλλη. Υπήρχαν ορισμένοι που μιλούσαν για τον νικέλιο κάδμιο τότε και άλλου οι οποίοι αναφέρονταν περισσότερο στο νικέλιο μέταλλο και στι ηλεκτρικέ στήλε που χρησιμοποιούν το υλικό αυτό. Και ήδη τότε ήταν δύο φορέ πιο αποτελεσματικό το νέο αυτό υλικό σε σχέση με τον νικέλιο κάδμιο και υπήρχαν τότε πολλοί εκπρόσωποι του βιομηχανικού κλάδου που μας λέγαν ότι οι στήλες νικελίου καδμίου ήταν πραγματικά απαραίτητες και ότι η ουσία αυτή έπρεπε να χρησιμοποιείται. Και τότε πριν από έξι χρόνια ουσιαστικά είχαν απευθυνθεί σε εμπειρογνώμονε στη Σουηδία που μου είχαν πει ότι δεν χρησιμοποιούμε προφανώ εμεί νικέλιο κάδμιο, αλλά λίθιο. Ήδη από το 2006 κάνουν αυτοί κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο να περιμένουμε λοιπόν τόσα πολλά χρόνια, δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να πρέπει να πάμε μέχρι το 2014, που ήδη είναι μια πολύ απομακρυσμένη χρονική προθεσμία. Δεν υπάρχει λόγο να περιμένουμε τόσο πολύ. Γιατί στην περίπτωση αυτή είναι περιττή και η ίδια η οδηγία η ίδια η αγορά θα προσαρμοστεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η οδηγία τελικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι για όλε αυτέ τι εφαρμογέ από περιβαλλοντική και αποτελεσματική πλευρά υπάρχει μια καλύτερη εναλλακτική λύση. Και είναι ψευδέστηση αυτή τη στιγμή να κάνουμε λόγο για ανακύκλωση κάθε φορά που μιλάμε για δράργυρο και νικέλιο δεν προβλέπεται ανακύκλωση του καδμίου, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε κάτι τέτοιο άλλωστε. Θέλουμε να εξαφανίσουμε, να εξαλείψουμε εντελώς την ουσία αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα γίνει τελικά είναι ότι το κάδμιο αυτό θα καταλήξει σε χωματερές. Θα πρέπει λοιπόν να εξαλειφθεί η ουσία αυτή το συντομότερο δυνατό γιατί όσο περισσότερο παραμένει η ουσία αυτή στην αγορά, ουσιαστικά εμείς ε, δημιουργούμε, συσσωρεύουμε τεράστιες ποσότητες καδμίου που ουσιαστικά θα φέρουν σε πάρα πολύ δυσμενή θέση τις μελλοντικές γενναίες. Προφανώς υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, όπως σας είπα, οι οποίες είναι και πολύ πιο αποτελεσματικές. Συμφωνώ επίση απόλυτα με τον εισηγητή όσον αφορά τα στοιχεία κουμπιά. Είναι πολύ θετικό ότι προσθέσετε το σημείο αυτό στην πρόταση. Και κυρία Κουκοβίτσε, Όντως υπάρχει μια ανάλυση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία λέει ότι είναι πολύ θετικό όντως το να εξαλειφθούν τα στοιχεία κουμπιά. Ήδη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε εξίσου φιλόδοξοι και με το χρονοδιάγραμμα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, απευθύνομαι σε εσά. Σα παρακαλώ πολύ, εφαρμόστε το άρθρο 11 και εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α φέρουμε την καταλεκτική ημερομηνία λίγο πιο νωρί. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ενδεχομένω μια διαφορετική όμω ημερομηνία για την απαγόρευση διάθεση στην αγορά και μια ξεχωριστή καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση τη ουσία αυτή από την ε, αγορά. Μια ξεχωριστή λοιπόν ημερομηνία για την απαγόρευση διάθεση στην αγορά και ενδεχομένω ένα χρόνο αργότερα να αποσυρθούν τα στοιχεία αυτά από την αγορά εντελώ. Η κυρία Βέστλοντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλά ήδη έχουν λεχθεί, λογικά και ενδιαφέροντα. Και όπως είπαν άλλοι συνάδελφοι, από το 2006 συζητάμε μια αναλυτικά, λύση για φορητά ηλεκτρικά μηχανήματα και μας είχαν πει τότε ότι δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είμαστε τώρα στο 2012 και ένα σημαντικό ποσοστό της ειδική αγοράς λειτουργεί με μπαταρίες που δεν περιέχουν κάδμιο. Οι εναλλακτικέ λύσεις, οι εναλλακτικέ μπαταρίες υπάρχουν, είναι λίγο ανταγωνιστικές και πρέπει αυτές τις μπαταρίες νικελίου, καδμίου να εξαφανιστούν. Έπρεπε να το είχαμε κάνει πριν από έξι χρόνια. Τώρα όμως είναι επίγον. Όσον αφορά τώρα τα, ε, τις μπαταρίες, τα στοιχεία κουμπιά με υδράργυρο, από ό,τι κατάλαβα η Κομισιόν έχει κάνει μία μελέτη και δείχνει ότι υπάρχουν και οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες να αντικατασταθούν αυτές οι μπαταρίες. Όσον αφορά ε, ο Ιδράγιος εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ακολουθήσει μία πολύ αυστηρή γραμμή για την ε, εξάλληψη του υδράργυρου και διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρουμε πόσο εξαιρετικά τοξικό είναι. Γιατί λοιπόν να υπάρχει μία ρήτρα εξαίρεση για αυτά τα στοιχεία κουμπιά με υδράργυρο είναι γεγονός ότι μπορούν, μπορούν να, ε, ε, να τα εξαλείψουμε τελείως, ε, να εξαφανιστούν από την αγορά και αυτό πρέπει να κάνουμε το ταχύτερο. Η Σοφία Κούνιχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Παναγιώτοφ για το εξαιρετικό του έργο για αυτή την αναθεώρηση τροποποίηση της οδηγίας διότι σκόπιμο και σημαντικό θα είναι να επιβάλλουμε στους πολίτες να αλλάξουν συνήθειες. Ιδίως παρεμβαίνοντας και ενισχύοντας το λίθιο σε αντίθεση με τον νικέλιο Κάδμιο. Για αυτό το λόγο νομίζω πολύ καλά εξισορρόπησε ο εισηγητής τις διαφορετικές παραμέτρους, ώστε πέραν του στοιχείου προστασία του πλανήτη, που είναι μια από τις βασικές μας μέρημνε, εξέτασε και τις οικονομικές πτυχές, κάτι που λόγω της συγκυρία οφείλουμε να συνεξετάζουμε. Λόγω χάρη θεώρησε ότι σκόπιμο είναι να παραταθεί κατά ένα έτος ή καταληκτική προθεσμία ώστε να προλάβει η αγορά να προσαρμοστεί. Να προλάβουν οι πολίτες να προσαρμοστούν το βρίσκω εύστοχο αυτό. Και θα ήθελα να του προτείνω και εγώ από την πλευρά μου, ίσως, να σκεφτεί κατά πόσον θα μπορούσαμε να πάμε και λίγο παραπέρα. Ιδίως στην αιτιολογική σκέψη 4 και το άρθρο, το πρώτο άρθρο, ως προς την ε, καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2016 μήπως θα μπορούσαμε να την παρατείνουμε κι άλλο, για τον εξής απλό λόγο. Σήμερα, κάποιοι πολίτες στα κράτη-μέλη έχουν αγοραστική δύναμη μικρότερη από τη δική μου, ε, ή του κυρίου Σλίτερ ή τη δική μου προσωπικά. Έχουμε συσσωρευτές ε, λιθίου και ηλεκτρικές στήλες λιθίου ακριβότερες από τις στήλες νικελίου καδμίου. Θα είχε λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε τι οικονομικό αντίκτυπο θα υπήρχε και για αυτούς τους πολίτες. Εάν από αλληλεγγύη και λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν θα μπορούσαμε να παρατείνουμε ακόμα ένα ή δύο έτη την ε, καταληκτική ημερομηνία. Ώστε να προλάβει το λίθιο να εδραιωθεί στην αγορά σε κάθε περίπτωση. Και έπειτα σε ό,τι αφορά το άρθρο 6 στην εδάφιο 3 προτείνεται σε επίπεδο εργαλείων εξοπλισμού που λειτουργούν με στήλες νικελίου καθμίου να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού. Αυτό δεν το βρίσκω σκόπιμο. Και αυτό γιατί θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε αλλαγή μόνον του σωρευτή ή της ηλεκτρικής στήλης. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα πρέπει να επεξεργαστούμε και επιπλέον απόβλητα. Θα έχουμε περισσότερη ανακύκλωση να κάνουμε. Ο εξοπλισμό δεν είναι αναγκαστικά όλο ε, άχρηστο και πρέπει να λαθεί. Θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε την υποχρέωση μετατροπή τη ηλεκτρική στήλη του συσσωρευτή. Αυτά τα δύο σημεία ήθελα να επισημάνω στον ε, εισηγητή. Αλλά όπω και εσεί και εγώ θέλω να συμβάλλω στην καλύτερη διαχείριση των πόρων, την βελτίωση της βιωτική, του βιωτικού επίπεδου, με τα προϊόντα όπως αυτά του λιθίου, που σίγουρα είναι προτιμότερα από τα προϊόντα νικηλίου καδμίου, αλλά όχι θυσιάζοντας το οικονομικό συμφέρον των ε, συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για το Καλ Σλίτερ να μιλήσει. Ναι, όντως. Αυτό δεν είναι ισχυρό επιχείρημα. 90% όλων των, ε, μηχανημάτων ε, so των Black and Decker όπως λέμε χρησιμοποιούν κάδμιο ε, χωρίς λόγο αν έχεις ένα σπίτι, καλύτερα είναι να έχεις... Ε, να μοιράζεσαι ε, τα φορητά αυτά εργαλεία με τους ε, γείτονες και τους άλλους συγκάτοικους παρά να έχει ο καθένας μία τέτοια φορητή συσκευή Black Decker στο σπίτι του με αυτές τις μπαταρίες. Ε, μισή ώρα θα τη χρησιμοποιήσουμε ας πούμε τη συσκευή αυτή για όλο τον κύκλο ζωής. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα ε, δεν ε, ισχύει για μένα, δεν με πείσει. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο να μοιραζόμαστε τη χρήση ενός μηχανήματος παρά να έχουν τέσσερις άνθρωποι ένα μηχάνημα και να είναι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Εντάξει, άμα έχω ανάγκη κάποιου Black and Decker, λέει ο πρόεδρο, θα πάω στον Κάρλ να μου το δώσει. Μάλιστα, γιατί όχι, λέει. Yes. Uh, ευχαριστώ, κύριε. Uh, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα μειωθούν οι μισθοί των ε, εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενδεχομένω για άλλους λόγους. Να αναφερθώ στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητή καταρχάς και στη συνέχεια θα απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα του Καρτ Σλάιτερ. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεσή του που ουσιαστικά υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την επιτροπολογία με τις κατεξοδότηση πράξεις με την διπλή νομική βάση που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική προκειμένου να φαίνεται ότι η ίδια η οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες βασίζεται στη νομική αυτή βάση που έχει να κάνει με την ιστορική αγορά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση είναι αρκετά φιλόδοξη, τουλάχιστον σε ένα τη σημείο, το ότι ε, προσθέτει και τα στοιχεία κουμπιά και συγκεκριμένα τον υδράργυρο στα στοιχεία αυτά. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε μετά την υποβολή της πρότασής μας και για αυτό το λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στην αρχική μας ανακοίνωση. Γίνεται λοιπόν μια σχεδόν πλήρης ανάλυση του αντικτύπου για την χρήση υδραργύρου στα στοιχεία κουμπιά και θα ληφθεί λοιπόν και αυτή η μελέτη υπόψη. Προφανώ αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη δική σα την προσέγγιση, θα πρέπει να δούμε έπειτα από κοινού τι θα κάνουμε με την πρόταση αυτή. Κάπου βέβαια που είστε λιγότερο ε, φιλόδοξος είναι η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπουμε εμεί για το 2015. Εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα χρόνο η καταληκτική αυτή ημερομηνία Εμείς βάσει της μελέτης αντικτύπου θεωρούμε ότι το 2015 είναι η καλύτερη καταληκτική ημερομηνία. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι στο Συμβούλιο οι οποίοι θέλουν μια περαιτέρω ακόμα παράταση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού θα καταλήξει η μεταξύ συζήτηση. Ενδεχομένω σε κάποια σημεία να είστε ακόμα πιο λεπτομερείς από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αφαίρεστε στην απόσυρση των υφιστάμενων αποθεμάτων και εξαρτημάτων από την αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τόσο λεπτομερή αναφορά, γιατί το θέμα είναι ότι έχουμε μία πρώτη διάθεση στην αγορά και έπειτα μπορούμε να έχουμε και μία δεύτερη, τρίτη διάθεση στην αγορά. Εσείς γίνεστε πολύ πιο συγκεκριμένο στη δική σας πρόταση, αναφέρεστε επίσης σε επιμέρους συσκευές, σε εξαρτήματα κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες στην ε, πρότασή σας, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο. Εφόσον βέβαια η πρότασή σας γίνει επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευθυγράμμιση επιτροπολογίας. Και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα τα δύο ζητήματα τα οποία έθιξε ο Καρλ Σλίτερ. Γίνανε διάφορες συναντήσεις, στις οποίες προσπαθούσαμε να δούμε ακριβώς τι γίνεται με το άρθρο 11. Αν δείτε το κείμενο της οδηγίας, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ουσιαστικά ένα πρόβλημα, το κείμενο της οδηγίας δεν είναι πάρα πολύ σαφές το σημείο αυτό. Λέω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί θα, θα σχεδιάζουν τις συσκευέ κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές να μπορούν να αφαιρεθούν δεν λέγεται από ποιον. Για ορισμένα κράτη-μέλη αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι παραγωγοί, οι κατασκευαστές είναι αυτοί που θα πρέπει να μπορούν να φέρουν τις μπαταρίες. Άλλοι πάλι πιστεύουν, άλλα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι αυτοί που θα μπορούν να φέρουν αυτές τις μπαταρίες από τις συσκευέ. Στην Τεχνική Επιτροπή που έχουμε με τη συμμετοχή των κρατών μελών συζητήσαμε το ζήτημα αυτό, τους είπαμε ότι θα το εξετάσουμε περαιτέρω στο μέλλον και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σαφή καθοδήγηση για το ζήτημα αυτό. Μα εγώ μίλησα με επαγγελματίε και μου είπαν ότι και αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να αφαιρέσουν αυτέ τι μπαταρίε. Καλό είναι να μην κάνουμε διάλογο. Είχατε ολοκληρώσει. Όχι απολύτω, αλλά σχεδόν. Θα εξετάσουμε λοιπόν περαιτέρω το ζήτημα αυτό και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αποσαφινιστεί πλήρως στα έγγραφα τα οποία θα δημοσιεύσουμε στο μέλλον. Πάντως, σας επαναλαμβάνω, το ζήτημα αυτό το συζητήσαμε πριν από ένα μήνα συγκεκριμένα με τα κράτη-μέλη. Μας απασχολεί λοιπόν και εμάς, δεν το έχουμε παραβλέψει. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την σήμανση. Υπάρχει κοινοτική νομοθεσία η οποία είχε εγκριθεί το 2010 όσον αφορά τις μπαταρίες εκείνες οι οποίες επαναφορτίζονται και έχει αρχίσει να ισχύει από το Μάιο του 2012. Από τεχνικής πλευράς είχαμε πρόβλημα με τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προσπαθούμε εδώ πέρα να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Αυτή τη στιγμή θα καταρτήσουμε το πρότυπο αυτό, το πρότυπο αυτό θα μας σε θέση να προτείνουμε και μία σχετική νομοθεσία. Το ζήτημα λοιπόν είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι προβλεπόταν στην αρχή και γι' αυτό το λόγο έχουμε καθυστερήσει. Δηλαδή έχουμε διαφορετικούς κανόνες σήμανσης για τις φορτιζόμενες μπαταρίες ενώ το, η κατάσταση είναι διαφορετική για τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και δίνω εν κατακλείδη το λόγο και πάλι στον εισηγητή. Ευχαρίστως. Ε, επεμβαίνω, παρεμβαίνω ξανά. Η συζήτηση αυτή ήταν πολύ ευχάριστη. Άκουσα με προσοχή όσους μίλησαν και θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα σε ερωτήσεις. Καταρχάς, να της κυρίας Κόκοβιτς. Την ευχαριστώ για τις πολύτιμες παρατηρήσεις της σε σχέση με τον Ιδράγυρο. Έχουμε ήδη ορισμένα αποτελέσματα. Μία έκθεση της Κομισιόν πέρσι για αυτό το θέμα. Η διαγραφόμενη τάση λοιπόν δείχνει ότι στις μπαταρίες δεν χρησιμοποιείται υδράργυρος ή όλο και λιγότερο και το 2013 θα γίνει ένας ε, ε, ενδελεχής διάλογος για αυτό το θέμα. Τώρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή να λυθεί το πρόβλημα του υδράργυρου. Απαντώντας ε, στον κύριο Σλούτερ, έθεσε πολύ σημαντικά ζητήματα και συμμερίζουμε απόλυτα τις απόψεις του. Όμως έκανα πάρα πολλές συζητήσεις με παραγωγούς, με καταναλωτές, με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους. Το κάδμιο πρέπει στα φωτοβολταϊκά και σε, ειδικές, ε, σε ειδικά υλικά να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το κάδμιο το οποίο συγκεντρώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και γι' αυτό είχαμε ζητήσει να μην χρησιμοποιούνται οι μπαταρίες νικελίου καδμίου. Βεβαίως έχουν, ελατώ, έχουν μειονεκτήματα αυτές οι μπαταρίες, χωρίς αμφιβολία. Χρειαζόμαστε λοιπόν καιρό διότι η βιομηχανία ανακύκλωσης δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα απόλυτα ικανοποιητικά και οι καινούριε μπαταρίες είναι ακριβές. Πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος έως ότου οι τιμές μειωθούν. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε και στο μέσο μιας οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά τα έχω αναλογιστεί, τα έχω σκεφτεί. Τώρα, εάν επιβάλλουμε απότομα την απαγόρευση θα ζημιωθούν με εκατομμύρια οι επιχειρήσεις διότι δεν είναι πρόθυμες ούτε έτοιμες να αλλάξουν την παραγωγή τους και να κάνουν μόνο καινούριε μπαταρίες. Το Ε, η πάυση χρησιμοποίησης ή μάλλον η επιβολή της απογόρευσης είτε είναι 2016 είτε 2020 θα γίνει. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω αυτή την διεύρυνση, την επέκταση για ένα χρόνο για να μπορέσουμε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2016 να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία προσαρμογής στους κατασκευαστές. Κύριε Γιώργη, σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας και σας υποστηρίζω. Συμφωνώ. Ε, εκεί που λέτε ότι το πρόβλημα με τις μπαταρίες ε, λυσίου είναι υπερβολικά ακριβές και επίσης έχουν προβλήματα επαναφόρτησης πολλά προβλήματα. Εάν δεν μπορούν να πως υπό συγκεκριμένε συνθήκες υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης να εκραγούν. Εκόμα, λοιπόν έχουμε τεχνικά προβλήματα με τις μπαταρίες λυθίου. Εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν που σε, μερικά, σε μερικές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης θα δημιουργηθεί μια κατάσταση απότεμος αλλαγής, ένα σοκ δηλαδή σημαντικό, διότι ξαφνικά θα υποχρεωθούν να παράγουν και να αγοράζουν μπαταρίες διπλού κόστους. Ευχαριστώ και την Επιτροπή, την Κομισιόν και τον εκπρόσωπο της ε, έχουν μια σωστή επιχειρηματολογία και έκρινα σωστά τους στόχους της έκθεσής μου. Ε, ευχαριστώ όλους όσοι συμμετέσχουν στη συζήτηση και η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Είχατε πει ότι θα υπάρξει μια γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής δεν υπάρχει αντίρρηση. Θα ζητήσουμε λοιπόν γνωμοδότηση από τη Γιούρη και η πρόθεσμια τροπολογιών είναι 5 ε, Δεκεμβρίου στις 23 ε, Ιανουαρίου θα συζητήσουμε το θέμα στην Επιτροπή και στις 19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και μάλλον θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Απριλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσοι, όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. 17 το οποίο είναι δικό μου θέμα, εγώ είμαι εισηγητής και πρόκειται για <laughs> τις οδηγίες πρωινού οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Καφέ, χώριο, σοκολάτα, διάφορα ζαχαροειδή, μαρμελάδες, κρεμοειδή και συμπυκνωμένου γαλακτός. δεν θα ήθελα τώρα, είδατε το γάλα που χύθηκε τις ε, τελευταίες μέρες με τις διαδηλώσεις εδώ στην πλατεία. Ο στόχος είναι να μπορέσει η Κομισιό να προσαρμοστεί στις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας και να ε, ε, καλύψουν, ε, ε, να δώσουμε την ευκαιρία στην Επιτροπή για να το κάνει αυτό, να διευρύνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες για αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στην Επιτροπή να μπορέσει γρήγορα να προσαρμόζει και να επικαιροποιεί τεχνικά στοιχεία σε αυτά τα παραρτήματα για να μπορεί να αποκριθεί στα σχετικά διεθνή πρότυπα. Η πρόταση επίσης λέει ότι θα ε, ακυρωθούν οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής εκεί όπου ήδη καλύπτονται από τις αντίστοιχες οδηγίες. πρέπει να πω ότι η πρόταση αυτή μέσα στα πλαίσια της επιτροπολογίας αντιπροσωπεύει ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προόδου. Δύο μόνος οδηγίες ε, παρουσιάστηκε αντίρρηση, κάποια αντίρρηση. Αυτό όμως πιστεύω ότι θα αλλάξει. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οδηγία για τα διατηρημένα γάλακτα ή ε, ολικά αφιδατωμένα γάλακτα έχει προσαρμοστεί όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες βάσει του κόντεξ αλιμεντάριους και εναρμονίζει την οδηγία με το πρότυπο του κόντεξ αλιμεντάριου σε αυτά τα προϊόντα. Ε, αυτή η οδηγία, εάν δώσουμε αυτές τις διευρυμένες εκτελεστικές αρμεδιότητες, θα μπορέσει να προσταρμοστεί γρήγορα μέσα στα πλαίσια ε, των ε, διεθνών συνθήκων. Η οδηγία για το, για τα φρούτα μοιάζει λοιπόν ε, με την οδηγία για τους χυμούς φρούτων 2012 κάθε 12 ε, όπου το παράρτημα το οποίο περιλάμβανε τις ονομασίε των προϊόντων εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής της ανάθεσης εξουσιών. Ε, γι' αυτό λοιπόν έχω επικεντρώσει αυτές τις εκτελεστικές αρμοδιότητες σε μη ουσιαστικά στοιχεία και ακολουθώ τη γραμμή ακριβώς ε, όπως εφαρμόστηκε στην τροποποίηση της οδηγίας για τους χυμούς φρούτων όπου η Κομισιόν επίσης θα λάβει αυτές ε, τις ε, εκτελεστικές αρμοδιότητες προτείνω τον περιορισμό της ανάθεσης εξουσιών σε μία ανανεώσιμη πενταετή περίοδο, καθώς και την παρακολούθηση της ανάθεσης των εξουσιών μέσω της υποχρέωσης της Επιτροπής να υποβάλει σχετική έκθεση πριν από τη λήξη κάθε πενταετούς περίοδου. Αυτά είχα να πω εν συντομία για τις οδηγίες πρωινού και την ε, προσαρμογή των εκκληστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ότι πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό έγγραφο αλλά πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί η νομοθεσία τα επόμενα χρόνια για όλα τα ζητήματα. Αναφερθήκατε στα εκχυλίσματα καφέ, στα εκχυλίσματα κυχορίου, στα προϊόντα κακάο και σοκολάτα, σε ορισμένα σάκχαρα, στι μαρμελάδες ζελέ, μαρμελάδε εσπυριδοειδών, κρέμα κάστανου κτλ. Όντως προσπαθούμε εδώ πέρα αγαπητοί συνάδελφοι να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου. Θεωρώ λοιπόν ότι τα στοιχεία των προϊόντων αυτών είναι πάρα πολύ σημαντικά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ενταχθούν στην διαδικασία κάτω εξουσιοδότησης. Οι συνομοθέτες θα πρέπει εδώ πέρα να συνεχίζουν να έχουν μία ενεργή παρουσία και να μην ανατεθούν όλα αυτά τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εναπόκειται λοιπόν στους συνομοθέτες να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό, καθότι δεν πρόκειται, δεν επίγει καθόλου το ζήτημα αυτό. Προφανώς δεν πρέπει να κλείσουμε την πόρτα στην καινοτομία ή στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας, αλλά παράλληλα δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία νομική αστάθεια. Σας υπενθυμίζω ότι οι επιχειρήσεις μας υποφέρουν από την νομική αυτή αστάθεια και πολλές φορές δεν καταφέρνουν ε, βραχυπρόθεσμα να χρησιμοποιήσουν ένα νομοθετικό μέσο όταν δεν ξέρουν πώς εξελίσσεται η κοινωνική νομοθεσία που τις αφορά. Συνοψίζοντα λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την τοποθέτησή του στην έκθεση αυτή. Σίγουρα πρόκειται για ένα ζήτημα τεχνικής φύσης, ένα εσωτερικό διοργανικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Αβώνας. παρόλα αυτά πρόκειται όμως και για ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον εισηγητή και είμαι στην απόλυτη διάθεσή του για μελλοντικέ ακόμα και διμερείς συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Σκιώδης, εισηγητής για τους φιλελεύθερους, είναι επόμενος ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας ανησυχεί να έχουμε να κάνουμε με τεχνικές εκθήσεις, αλλά βεβαίως η ευθυγράμμιση με, συνθήκη της, με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι πάντοτε κάτι που το βρίσκουμε υποφελές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν εδώ πώς ε, θα ορίσουμε τις αρμοδιότητες και ποιο θεσμικό όργανο θα τις αναλαμβάνει. Επίσης, πρέπει να ορίσουμε και πού τοποθετούμαστε εδώ σε σχέση με την αρχή της επικορικότητας. Έχουν τόση καχυποψία για την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οι πολίτες. Θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς η Ένωση να πάει κοντά στους πολίτε. Και αυτό θα το πετύχουμε σε όλη τη διαδικασία την νομοθετική, εφόσον αυτή είναι συνεπής. Και υπάρχει περιθώριο οι πολίτες να μπορούν να εκφραστούν και εκείνοι σε κάποιο βαθμό. Τώρα, για το εύρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και αν θα πρέπει να σκέφτονται την επικαιροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών τα κράτη-μέλη ή το Κοινοβούλιο, εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένε οδηγίες που είναι αρκετά απερχαιωμένες. και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να δούμε πόσο συχνά έχουν ε, μεταβληθεί, γιατί και πώς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον ήταν μια θεωρητική προσπάθεια ή ανταποκρινόταν σε εξελίξεις που ήδη λάβαιναν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτά πώς μπορούν να προσαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ στο Κοινοβούλιο θυμάμαι πριν από δύο χρόνια είχαμε μια ολόκληρη διαφιλονικία για το πώς θα ορίσουμε τη σοκολάτα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναρωτιόταν αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σοκολάτα τύπου Βρετανικού. Το κακάο, ας πούμε, με το οποίο φτιάχνουμε ζεστή σοκολάτα. Θυμάμαι πρώην συναδέλφου, τον κύριο Γκάλαχερ, ε, πρώτο σελίδα στι εφημερίδε. Φαίνονται πολύ τεχνοκρατικά όλα αυτά και γραφειοτικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία. Πρόεδρε, εδώ θα πρέπει να έχουμε κατακρισοδότες πράξη, διότι θέλουμε ακριβώ να ανταποκρίνονται, να απηχούνται και οι εθνικέ ευαισθησίε σε τόσο τεχνικές σε τόσο τεχνικά νομοθετήματα. Για τη μαρμελάδα, α πούμε. Τι μπορεί κανεί να προσθέσει στη μαρμελάδα. Ποια είναι τα συστατικά μια σωστή μαρμελάδας. Θα μπορούσε όντω να αναλάβει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί κάποιο να θέλει να προσθέσει κάτι τελείως ακίνδυνο. Αλλά τα χαρακτηριστικά της μαρμελάδας να μεταβάλλονται όντως. Εδώ λοιπόν, Πρόεδρε, ε, προτείνεται διαγραφή του παραρτήματος 2 από την προτάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θα υπάρχει αλλαγή εδώ στο παράρτημα 2, θα επηρεάζεται το παράρτημα 2. Όμω, εγώ έχω και την εξή αμφιβολία. Θα επηρεαστεί η ποιότητα των τροφίμων μα. Ε, με το παράρτημα 2 αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της μαρμελάδας, όπως είπα. Μπορεί κάτι να προσθεθεί και χωρίς κάτι άλλο να αφαιρεθεί, αλλά να αλλάζει ο χαρακτήρας της μαρμελάδας. Λοιπόν, είναι σημαντική η έκθεση, παρόλο που φαίνεται τελείω τεχνική και θα πρέπει να το δούμε με προσοχή, εάν όντω πρέπει να γίνει αυτή η διαγραφή, όχι και το καθεξή. Ευχαριστώ. ως πρόεδρος ε, διατύπωσε έτσι την έκθεση όπως μπορούσα καλύτερα. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά θα, θα πω εγώ τον τελευταίο λόγο. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο έκθεσης. Προφανώς εμείς ε, υπερασπιζόμαστε την δική μας την πρόταση, τη δική μας τη γραμμή που βλέπετε στην ανακοίνωσή μας, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις ε, κατεξοδότηση πράξεις προκειμένου να τροποποιούμε κάποιες παραμέτρους. Εσείς στην ε, έκθεσή σας και στην εισαγωγή του κειμένου αναφέρεστε επίσης και στην οδηγία για τους χυμούς φρούτων και κάνετε ένα παραλληλισμό. Στην οδηγία όμως αυτή έχουμε άλλους ορισμούς, τι είναι νέκταρ, τι είναι χυμός φρούτου, και έχουμε όμως τεχνικές παραμέτρους που είναι σε ένα άλλο παράρτημα που μπορεί να τροποποιηθεί με πράξεις εξοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ τώρα όλες οι παράμετροι και οι ορισμοί στο κείμενο βρίσκονται στην, στο ίδιο τμήμα πλέον. Δεν ξέρω λοιπόν σε ποιο βαθμό θα καταφέρουμε να δικαιολογήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο στο μέλλον το ότι έχουμε μία πολύ δαπανηρή νομοθετική διαδικασία προκειμένου να καταφέρουμε να τροποποιήσουμε κάποιες πολύ τεχνικές συσκευές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιες πολύ συγκεκριμένες ουσίες. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα καταφέρουμε να δικαιολογήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο το ότι τελικά επιθυμούμε εσείς, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εγκρίνεται μια πολύ δαπανηρή διαδικασία και βραδύ διαδικασία για να γίνει μια τροποποίηση του εν λόγω κειμένου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράιμανς έχει κάτι να ρωτήσει. Α, ρώτησε κάτι και δεν απαντήσατε νομίζω ή όχι, κάνω λάθος. Es um Πρόκειται για τον ορισμό, ήταν το ερώτημα δηλαδή, αν η Κομισιόν έχει ήδη παρέμβει ή όχι. Η, κυρία, η συνάλφος κυρία Ράιμας για... Ε, ε, έθεσε το ερώτημα και πόσες φορές έχει ε, χρειαστεί τα τελευταία χρόνια να παρέμβεται η Κομισιόν για τον ορισμό εξαρτάται εάν στον ορισμό περιλάβει κανείς και τις παραμέτρους. Για τον ίδιο τον ορισμό αυτό καθεαυτό μία φορά έγινε μία αλλαγή, αλλά για τις παραμέτρους μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν πολύ πιο γρήγορα, ανάλογα με τις τεχνικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Και γενικά αυτό που συνέβη στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι θα αναλυφθεί και στο μέλλον. Οι τεχνικές ε, εξελίξεις προχωράν πολύ γρήγορα και πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αλλάξουν αυτές τις παραμέτρους. Ε, σύντομα. Ξαναρωτάω, λέει ο πρόεδρος, υπήρξε στο παρελθόν η ανάγκη μίας παρέμβασης της Κομισιόν χρειάστηκε να αλλάξετε, να παρέμβετε γιατί χρειάζεστε ακριβώς αυτές τις εκτελεστικές αρμοδιότητες η Κομισιόν. Εάν ε, αναφέρεστε στο επιχείρημα ότι αυτές οι αλλαγές δεν θα γίνονται συχνά, συμφωνώ. Όμως το θέμα είναι τη μία φορά που θα χρειάζονται μπορούμε να τις κάνουμε. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα γίνονται συχνά. Δεν είναι ο χρόνος το καθοριστικό επιχείρημα. Απλώς δεν θα έχουμε την αναγκαία διαδικασία να αλλάξουμε μία τεχνική λεπτομέρεια και θα καθυστερήσουμε με μία χρονοφόρο διαδικασία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα μπορούσατε ίσως να μας ε, ενημερώσετε γραπτός πόσες φορές ε, χρειάστηκε αυτή η χρονοβόρη διαδικασία να παρέμβεται, ποιο ήταν το κόστος που αναφέρεται το υψηλό κόστος στους φορολογούμενους. Πάντως, σας ευχαριστώ όλους για την συμβολή σας στη συζήτηση και για αυτά που είπε η Λίντα Μακέβαν. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει σαφώς να δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ταχύτερο δυνατόν όταν ε, είναι η ανάγκη, όταν πρέπει να κάνουν αυτές τις τεχνικές αλλαγές. Το, τα δικαιώματα τα οποία κερδίσαμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει και να τα υλοποιήσουμε. Δεν θέλουμε μία αύξηση ε, κόστους ε, και αύξηση των δαπανών. Πρέπει να είμαστε ε, να έχουμε μία ευελιξία για να μπορούμε να προσαρμοστούμε γρήγορα, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατία και κόστος. Αυτό πρόκειται λοιπόν για μία προσαρμογή. προσαρμογή για να μπορέσουμε γρήγορα να εφαρμόσουμε το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας θα γίνει μία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Θα οργανωθεί για να συντονίσουμε τις θέσεις μας και η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 5 Δεκεμβρίου στις 23 Ιανουαρίου μαζί με τις τροπολογίες θα συζητήσουμε το θέμα και υποθέτω στις 19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Απριλίου του χρόνου. Στην ημερήσια διάταξη. Φτάσαμε στο τέλος της ημερησίας διάταξής μας. Αύριο θα αρχίσουμε στις 10. Έχουμε τον κύριο Ντάνσετ, εκτελεστικό διευθυντή Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Όλοι οι συνάδελφοι είναι προσκεκλημένοι και θα ήθελα το, τα στελέχη μας να φροντίσουν να ε, φέρουν όσο περισσότερο σε ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Επίσης, χαιρετίζω θερμά, γιατί το είπα και το πρωί, τους 8 δημοσιογράφους οι οποίοι ήρθαν μετά από πρόσκληση της συναδέλφου Χίμπνερ. Σας καλωσορίζω και ελπίζω να αποκομίσετε ε, μια καλή εντύπωση από τις εργασίες μας. Σας καλωσορίζω και αντίο.